Τη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα. Περιμένουμε την ε, κυρία Επίτροπο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων την κυρία Εσλέρ Μπεγκίν, η οποία σε τέσσερα λεπτά θα μας εξηγήσει το πρόβλημα. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών που είχε την ευγενή καλοσύνη να δεχτεί τη διαδικασία το άρθρο 91, το κατεπήγον αυτό ψήφισμα δηλαδή, γιατί και στην προηγούμενη μας ολομέλεια είχαμε ένα κατεπήγον ψήφισμα για το ίδιο θέμα του, της Σρι Λάνκας. Και ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο που δέχτηκε να ξαναγίνει αυτή η συζήτηση και ευχαριστώ και εσάς κυρία Επίτροπε που προσήλθατε σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Θελήσαμε όμως να κάνουμε μια πολιτική χειρονομία και να δώσουμε ένα μήνυμα στους εκπροσώπους και της κυβέρνησης και του κινήματος των Ταμούλ γιατί η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Έχουμε μαρτυρίες από οικογένειες Ταμούλ που βρίσκονται στην Ευρώπη και που συνεχώς μας στέλνουν μηνύματα και μαρτυρίες για αυτά που συμβαίνουν εκεί στις οικογένειές τους που έχουν παγιδευτεί στις διαμάχες μεταξύ των τίγρεων του Ταμούλ και των δυνάμεων της κυβέρνησης της Σριλάνκα. Δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι οι παγιδευμένοι, αλλά υπολογίζουμε μεταξύ 150 και 200 χιλιάδες. Οι άνθρωποι αυτοί ζητούν να κενωθούν από τις εμπόλεμες περιοχές. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις λένε ότι η εκένωση αυτή μπορεί να γίνει δια θαλάσσης, αλλά πού θα πάνε έστω και δια θαλάσσης. Το απόγευμα γνώρισα μία κοπέλα που γεννήθηκε σε στρατόπεδο προσφύγων στη Στριλάνκα και ζει σήμερα στην Ευρώπη και ξέρω ότι αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί να ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων. Δεν είναι ούτε αυτό λύση. Ζητούμε λοιπόν στο ψήφισμά μας να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός. Έγινε συζήτηση με το ΕΛΚ για το κατά πόσο πρέπει να είναι μόνιμη ή προσωρινή η εκεχηρία αυτή. Πάντως ζητούμε κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουν οι πληθυσμοί αυτοί να φύγουν. Και βέβαια ζητούμε επίσης στο ψήφισμα η κυβέρνηση της Σριλάνκα να συνεργαστεί με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με τις χώρες που ζητούν την επίλυση της διαμάχης. Επίσης θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει να μεταφερθούν εκεί τρόφιμα και φάρμακα. Και τέλος, αν μου το επιτρέπετε, εξ ονόματος της ομάδας μου, γιατί με πρωτοβουλία των Πρασίνων καταθέσαμε αυτό το κατεπήγον ψήφισμα τη Δευτέρα στην Επιτροπή Εξωτερικών. Ζητούμε λοιπόν το θέμα να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους συναδέλφους που έχουν συμφέροντα στη χώρα αυτήν Μερικές πολιτικές ομάδες ζητούν εδώ και καιρό να συζητηθεί το θέμα της Σριλάνκα αλλά για εσωτερικούς λόγους ορισμένων ομάδων δεν μπόρεσε να συζητηθεί ούτε το θέμα των Ταμούλ και της κατάστασής τους, ούτε το θέμα της Σριλάνκα γενικότερα που το πρόβλημα υπάρχει από τη δεκαετία του 80 ήδη. Εφόσον είστε εδώ λοιπόν κυρία Επίτροπε θα ήθελα να θέσω και ένα πρόσθετο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα να επιλύσει ορισμένες διαμάχες και σειράξεις. Ίσως είναι λοιπόν ευκαιρία και τώρα και σήμερα να δούμε αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί εδώ μια μονάδα επίλυσης διαμαχών ή σειράξεων γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνεται σοβαρά υπόψη διεθνώς με τις προτάσεις που κάνει και δεν πρέπει να παραμείνει απλώς θεατής αλλά να προωθεί όντως την επίτευξη λύσεων στις σειράξεις. Και αν σήμερα μπορεί το ψήφισμα αυτό να αποτελέσει μια πρώτη τέτοια χειρονομία και αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα για τους ενδιαφερόμενους νομίζω ότι θα έχει ωφεληθεί πολύ η κοινότητα, η Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Και τώρα η κυρία Επίτροπος Φεραίρο Βάουμπνερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, δεχτώ την κυρία Ισλερβεγγιά. Σαν ε, ένα συμπρόδρο τη ε, διαδικασία ειρηνευτή του Σρι στο Τόκιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ κοντά τι εξελίξει στο Σρι και πραγματικά ανησυχούμε εντονότατα όσον αφορά την κατάσταση σήμερα και τις τραγικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις της διαμάχης αυτής όπως εκφράζεται και στα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις 27 Φεβρουαρίου και η δήλωση αυτή του Κομισιόν που έγινε επί τόπου από τους Συμπροέδρους ήταν της 3ης Φεβρουαρίου και έλεγε τα ίδια πράγματα. Έχουμε επίσης τους εκτοπισμένους που έχουν ε, ε από τις ε, μάχες στη Βόρεια στη Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μία κρίση, έχουμε μία ανθρωπιστική καταστροφή. Mm. Μας το επιβεβαίωσαν αυτό πολλές ανεξάρτητες πηγές συμπεριλαμβανομένου του ΟΕ και του Διεθνούς Ρητρού Σταυρού. Η κυβέρνηση πρότεινε ότι θα άνοιξε δύο δρόμους ε, για την διαφυγή των ανθρώπων αυτών. Αυτό μου είναι θετικό καταρχήν, αλλά στην πράξη τι θα γίνει. Κάναμε έκκληση σε όλα τα μέλη, στους αρχές της Ριλάνκα, αλλά και στους ε, τίγρης και σε άλλους για να προστατεύσουν τον ε, άμαχο πληθυσμό όπως προβλέπεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να τους επιτρέψουμε να εγκατασταθούν αλλού και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η LTT και ο Νιγηριανός στρατός είναι υπεύθυνοι για ζωτάς αριθμούς θυμάτων μεταξύ των αμάχων τους τελευταίους μέρες. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται κατά ανάγκη να δράσουν για να σώσουν ζωές στη Σρι Λάγκα πράγμα που επιβεβαιώθηκε από τον κύριο Τζον Χόλμ. τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Επίσης τέτοια είπε και το Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Όλα αυτά θα έχουν μόνιμες επιπτώσεις στην ειρήνη, στην συμφιλίωση και το μέλλον του Σρι και γι' αυτό υποστηρίζουμε ε, αυτά που είπε ο Σερ Τζον Χολ προς την κυβέρνηση του Σουράντα να διακόπουν οι εχθροπραξίες να επιτραπεί στους άμαχους πληθυσμού να φύγουν και να συμφωνήσουν σε μια ειρηνευτική διακοπή και ε, περάτωση των ε, ε, των ε, εχθροπραξιών. Δυστυχώς αυτή η έκκληση όμως αγνοήθηκε. Απορρίφθηκε. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση του, της Σρι έχει υποχρέωση να προστατεύσει όλους τους, τους πολίτες, όπως λέγεται και θα συμπεράσματα του Συμβουλίου τελευταία φορά, για να μπορέσουν οι άρρωστοι, οι τραυματισμένοι να φύγουν από εκεί και να τους επιτρέψουν να λάβουν φάρμακα και τρόφιμα. Αυτό το πρότεινε και η Ινδία την περασμένη εβδομάδα, περασμένο Σαββατοκυριακό. Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική. Και υπάρχουν επίσης απαγωγές, ε, θανατώσεις ε, και απειλές κατά των ΜΜΕ. Και εν όψη όλων αυτών θα πρέπει η, Κομισιό, ε, το, κυβέρνηση να διώξει τις πιο εμφανείς ε, περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει α, κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει μία στρατιωτική λύση στις εθνοτικές ε, διαμάχες, στα εθνοτικά προβλήματα της Σρι η μόνιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που οδήγησαν στην εξέργηση αυτή στην αρχή και να υπάρχει σωστός χώρος για τις δύο κοινωνίες. Και εγώ συμπρόεδρος πάντα είπα ότι μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να οδηγήσει σε μια ε, μόνιμη λύση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τη συζήτηση λοιπόν. Να ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Εξ ονόματος του ΕΛΚ για δύο λεπτά ο Τσάρλ Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η βάναυση εμφύλια σύρρηξη της Σρι Λάνκα πλησιάζει προς το τέλος, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει αυτό για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες ε, και τους τίγρης δεν ξέρουμε κατά πόσον θα δοθεί η δυνατότητα στους τίγρεις να, να διοργανωθούν και ίσως να χάσουν τελικά με περισσότερα θύματα. Αν υπάρξει μακροπρόθεσμη πάυση ψηρό, πυρός ε, θα υπάρξουν προβλήματα διότι ε, τα πρόσφατα γεγονότα αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι είναι ανελαίτη και ματοδιψής και ε, θα πρέπει να υποστηρίξει ο πρόεδρος τη λήξη μιας ε, σύραξης η οποία οδήγησε τη Σρι σε μια ε, πάρα πολύ μεγάλη και δυσχερή, δυστυχία και δυσχερή κατάσταση σε αυτό το όμορφο νησί. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φύγουν για να μπορέσει ο στρατός να ολοκληρώσει την ε, επίθεσή του. Δυστυχώς οι τίγρεις εκμεταλλεύονται τους ε, πολίτες ε, και τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες. Η διεθνή κοινότητα τους παρακινεί να παρετηθούν και να δημιουργηθεί και μια κατάλληλη δίωδος διαφυγής. Θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη δίωδος διαφυγής από, για τους αθώους πολίτες από την ε, περιοχή της σύραξης για να μπορέσουμε να αποφύγουμε χειρότερα πράγματα. Δυστυχώς ε, η υπομονή του στρατού είναι περιορισμένη και η φόβη ότι οι τίγρες θα προσπαθήσουν να διαφύγουν δια ε, ε, με τους αθώους πολίτες ε, ε, είναι υπαρκτή. Γι' αυτό εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητάμε να δημιουργηθεί ένας ανθρωπιστικός διάδρομος για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να διαφύγουν αλλά ζητάμε επίσης και μία ειρηνική δίκαιη λύση για για μια μουλτιεθνική Σρι Λάνκα, ώστε να υπάρχει και αξιότιμη, αξιότιμος καταμερισμός των πόρων και ειρηνική διαβίωση στη Σρι Λάνκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Ρόμπερτ Εύανς, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση και την παρουσία της Επιτρόπου, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ σοβαρή και ε, εις βάθος δήλωσή της. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Είναι κρίμα που το συζητάμε στις 11 η ώρα τη νύχτα με τόσο λίγο κόσμο, αλλά η παρακολούθηση δεν αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, ούτε το πώς νιώθουν πολλά από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Όπως είπε και η ίδια η Επίτροπος, ε, ανησυχούμε βαθύτατα για την κατάσταση και η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι η κατάσταση έχει προχωρήσει και όπως είπε και η κυρία Έσλερ στην αρχή, θα πρέπει να αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα για την επιδεινούμενη κατάσταση κατάσταση ε, η οποία όλο ένα και επιδεινώνεται περισσότερο κάθε μέρα. Υποστηρίζω το ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε με την εξαίρεση του όρου temporary, προσωρινός. Ο κύριος Τάνοκ ε, είπε ότι η μακροχρόνια κατάσπαυση πυρός ε, θα αποβεί καταστροφική. Ε, δεν ζητάμε μόνο προσωρινή κατάπαυση πυρός. Ε, οπουδήποτε υπάρχει σύρεξη ανά τον κόσμο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζητά πάντα μόνιμη κατάπαυση πυρός. Μια μόνιμη κατάπαυση πυρός η οποία θα ανοίξει το δρόμο, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για διπλωματική ανασυγκρότηση, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ο διάλογος και όντως να έχουμε αυτό το, την ειρηνική δίκαιη και πολυεθνική κοινωνία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τάνοκ και με την οποία συμφωνώ. Υποστηρίζω λοιπόν τους πρασίνους για την πρώτη του τροπολογία, την υπαριθμόν 1 και πιστεύω ότι οποιοδήποτε είναι αξιοπρεπής εδώ ανησυχεί για τους αθώους πολίτες στη ε, Σρι Λάνκα. Η προσωρινή κατάπαυση πυρών εξορισμού σημαίνει ότι θα επανέλθουμε στον πόλεμο αργότερο, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, η επιστροφή στον πόλεμο σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερους θανάτους, περισσότερο πόνο και περισσότερες ανθρωπιστικές δυστυχίε. Και δεν πιστεύω ότι κανείς εδώ ε, σε όλες τα έδρανα της Ολομέλειας, δεν το επιθυμεί αυτό. Η τροπολογία 2 καταδικάζει οποιαδήποτε πράξη βίας ε, από οποιονδήποτε και το κάνει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία περίπτωση βίας, ακόμα και τις πρόσφατες ε, επιθέσεις αυτοκτονίας που αναφέρθησαν. Να περάσω τώρα στις τροπολογίε 3, 4 και 5 και αν μου επιτρέπετε αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να διαβάσω ένα σύντομο κείμενο το οποίο έλαβα από ε, κάποιον βουλευτή στη Σρι Λάνκα, τον κύριο Σλα... Σάλβαρας ε, με ημερομηνία 8 Μαρτίου. Θα ήθελα να επισημάνω τους θανάτους ε, από τους ε, από το στρατό του Σρι Λάνκα ε, μεταξύ 8 και 10 στην ε, Τρίτη στις 10 Μαρτίου μεταξύ 8 ε, και 10 το πρωί. Χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρες φέρες, πολλές από αυτές είναι απογορευμένες σε πολλές χώρες. Πάνω από 130 πολίτες σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά. Κανένας δεν θα μπορούσε να ε, προτείνει ότι αυτά είναι κατασκευασμένο δημοσίευμα και προτείνω να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να συνδράμουμε και να λήξει αυτή η βία. Ο κύριος Κανακαταράκνουμ, ο οποίος ζει ε, εν μέσω της ε, περιοχής η οποία καλείται ασφαλής, είπε ότι από τις 2 Μαρτίου σήμερα 200 44 άτομα σκοτώθηκαν από βομβιστικές επιθέσεις και ε, είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς λέμε, ε, λέγεται ότι υπήρχαν βομβαρδισμοί από αέρος που σκοτώνουν περίπου 30-40 άτομα ημερησίω. Δεν πιστεύω, συνάδελφοι, ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει τέτοια δημοσιεύματα. Ε, από όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όλα τα στοιχεία που έχουμε από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, φαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Η τροπολογία 6 αναφέρεται ε, να σταθώ στην έκθεση του Σερ Τζον Χόλς την οποία μα έστειλε ο πρεσβευτή των Βρυξελών στη Σρι και παραθέτω ότι υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλά άτομα, υπάρχει υπερπληθυσμός και στα προσφυγικά στρατόπεδα και υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Έχω κάποιες φωτογραφίες, μου εστάλησαν ε, και εγώ πιστεύω ότι είναι αυθεντικές, δεν είναι παραποιημένες και νομίζω ότι η βοηθός της Επιτρόπου παρακολουθεί ε, τις εξελίξεις Επιτόπου και ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην επικίνδυνη ζώνη. Στην τροπολογία 7, 8 και 9 ε, θεωρώ ότι ενισχύουν την αρχική δήλωση στην εμπόλεμη ζώνη ώστε να μπορέσουμε να φροντίσουμε ε, τους αθώους πολίτες. Ζητάμε να υπάρχει πρόσβαση στην ε, περιοχή της μάχης αλλά και στα προσφυγικά στρατόπεδα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό το υποστηρίζει όλη η Ολομέλεια. Όλοι εδώ υποστηρίζουμε την βοήθεια των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Και τέλος θα πρέπει να γίνει κάτι και από πλευρά Ηνωμένων Εθνών, διότι πιστεύω ότι πρόκειται για μια διεθνή ανθρωπιστική κρίση, το λέει και ο ίδιο ο τίτλο, γι' αυτό και ακριβώ ευχαριστώ του πρασίνου που κατέθεσαν ε, το σχετικό ψήφισμα και ε, θα ήθελα να υποστηρίξω όλε τι τροπολογίε που κατέθεσαν όλε οι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ισλερ Μπεγκίν, εξ ονόματος των Πρασίνων, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ξανά την κυρία Φεραίρο Βάλτνερ για αυτά που μας είπε και για την ανταπόκριση που έδειξε στο αίτημά μας για βοήθεια στους πληθυσμούς αυτούς. Πράγματι φοβόμαστε μήπως αντιμετωπίσουμε παρόμοια κατάσταση όπως στη Βυρμανία το 2006 οπότε και η Χούντα εκεί είχε εμποδίσει την έξοδο των πληθυσμών από τις εμπόλεμες περιοχές. Θέλω όμως να απευθυνθώ και στους συναδέλφους εδώ του ΕΛΚ και των σοσιαλιστών διότι νομίζω ότι πρέπει κύριοι συνάδελφοι να επιδείξουμε κάποια φρόνηση εδώ. Το ψήφισμα το κατεπήγον ψήφισμα το καταθέσαμε για να εκφραστεί το κοινοβούλιο, να έχει αύριο μία θέση. Δεν θέλω όμως σε καμία περίπτωση για λόγους πολιτικών διαφορών που τις κατανοούμε γιατί τα έχουμε ξαναπεί για την άμεση, μόνιμη ή προσωρινή εγκεχηρία. δεν θα θέλαμε να καταψηφιστεί για αυτούς τους λόγους το ψήφισμα. Θέλω να πω όμως ιδιαίτερα προς τον κύριο Τάνοκ ότι επαναλαμβάνω με τα ίδια τα λόγια της Επιτρόπου καμία ένοπλη σύραξη δεν έχει ποτέ λύσει κανένα πρόβλημα. Αυτό το ξέρουμε. Ο πόλεμος ποτέ δεν λύνει τα προβλήματα. Το να ζητάμε λοιπόν μία προσωρινή εκεχηρία νομίζω ότι δεν είναι υπεύθυνη στάση προς τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς. Δηλαδή προβλέπουμε στο μέλλον να ξαναρχίσει πόλεμος, πότε δηλαδή. Όποτε έχει εκενωθεί ο πληθυσμός και πότε θα το ξέρουμε, μπορούμε να περιμένουμε. Οι Ταμούλ είναι οι ιδιοκτήτες της γης αυτής, είναι ντόπιοι, δεν είναι ξένοι κατακτητές. Μπορώ όμως να κάνω υποχωρήσεις και να αποσύρω τροπολογίες εάν πρόκειται όμως από κοινού αύριο να έχουμε την ίδια θέση για να δώσουμε αυτό το πολιτικό μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Τελείωσαν εδώ οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Τώρα οι λοιποί βουλευτέ. Πρώτα πρώτα ο κύριος Φανόρντεν για τρία ολόκληρα λεπτά. Δεν έχω καμία αυταπάτη για τις τρομερές επιπτώσεις του πολέμου στους αμάχους και θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγκρίναμε το προηγούμενο κατεπήγον ψήφισμα πριν από τρεις εβδομάδες για τη Σρι Εδώ και δεκαετίες η Σρι Λάνκα υφίσταται μια τρομοκρατική καμπάνια με οδηγούς τους τίγρης των Ταμούλ και κατά των δημοκρατικών κυβερνητικών δυνάμεων. Γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις αυτοκτονίας, χρησιμοποιούνται παιδιά ως στρατιώτες και τα τελευταία 26 χρόνια έχουν γίνει χιλιάδες δολοφονίες, πρόσφατα 40 θύματα κατά τον εορτασμό μιας Ισλαμικής ε, σε τέτοιες περιπτώσεις οι δράστες όπως οι τίγρες του Ταμούλ στρέφονται προς τον διεθνή παράγοντα. Ελάχιστα μέλη του κοινοβουλίου μας εδώ δυσαρεστήθηκαν από το ψήφισμα της προηγούμενης φοράς και ήθελαν και τότε να καταδικάσουν την κυβέρνηση της Σριλάνκα. Δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε τροπολογίες που βασίζονται σε φήμες και μάλιστα ανεπιβεβαίωτες ή επιλεκτικές αναφορές σε δηλώσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτά που μας λέει η κυβέρνηση. Πριν από έξι μέρες κύριε Πρόεδρε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε από τους τίγρεις να αφοπλιστούν και να εκενώσουν τους αμάχους και να συνεργαστούν με όλες τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη δράση των τίγρεων που εμποδίζουν την εκένωση των αμάχων. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να ζητήσουμε από τους τίγρεις να καταθέσουν τα όπλα και να απελευθερώσουν εκεί τους αμάχους η ανθρωπιστική βοήθεια τότε θα μπορέσει να χορηγηθεί και θα μπορέσουν να ελπίσουν επιτέλους σε μια ανθρώπινη ζωή οι πληθυσμοί αυτοί. Μόνο έτσι με δημοκρατικό τρόπο θα μπορέσει να οικοδομηθεί μια ευημερούσα κοινωνία για όλους τους πολίτες χωρίς την τρομοκρατική καταπίεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κ. Τζολάινεν. Κύριε συμφωνώ πολύ μαζί σας ότι ε, χρειάζεται μια πολιτική και όχι μια στρατιωτική λύση στη Σρι Λάγκα. Ήμουν πολλές φορές στην χώρα αυτή σαν μέλος της αντιπροσωπείας ε, με την ε, Σρι Λάγκα και ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί μετά από 25 ετών βία. Δεν θα σας πω βέβαια όμω ότι σε ένα τέτοιο πόλεμο θα πρέπει οι τίγρες του Ταμούλα κάνουν κάποια βήματα που δεν τα έχουν κάνει Είπατε και εσείς ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών στις 23 Φεβρουαρίου κάλεσαν έντονα την οργάνωση αυτή να καταθέσει τα όπλα. Για φανταστείτε μια χώρα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να υπάρχει από 25 χρόνια ε, τρομοκρατία. Πολλά είναι χαόδηση στην περίπτωση αυτή. Μπορεί κανένα εύκολο να το φανταστεί. Εγώ είμαι υπέρ των προβλημάτων των Ταμούλ. Από την μεριά μου φαίνεται βέβαια ότι είναι αδύνατο να παραβλέψουμε την άλλη πλευρά. Υπάρχουν ε, εκατοντάδες χιλιάδων, ε, χιλιάδες άτομα σε αυτό το μικρό τη μικρή ζώνη και μάλιστα σήμερα υπάρχει και μία δήλωση στον τύπο ότι σύμφωνα με όσα είπαν οι μάρτυρες ε, πυροβολούνται εκείνοι που θέλουν να φύγουν από τη ε, ζώνη αυτή. Και θα πρέπει αυτές οι πρακτικές να σταματήσουν, να τελειώσουν. Δεν επιτρέπεται να συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. Γιατί ο ομοσπονδισμός βρίσκεται ανάμεσα στα και των δύο πλευρών και θα πρέπει να κάνουμε βέβαια και μία έκκληση προς την κυβέρνηση να επιτρέψει ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό θέμα και από τις δύο πλευρές ε, και θα πρέπει νομίζω να προετοιμαστούμε για το τι θα γίνει μετά το πόλεμο. Το είπατε εσείς και μετά ότι το 13ο, η 13η τροπολογία του συντάγματος του Σρι θα πρέπει να σχετίζεται με κάποια μέτρα για τους πληθυσμούς που ζουν εκεί. Εκεί μπορεί να βοηθήσει η Κομισιόν και είμαι σίγουρος ότι εσείς στην Επιτροπή και εμείς στο Κοινοβούλιο θα βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Περνάμε στο ΚΑΤΣΙΑΙ. Ο κύριος Ρούμπ το λόγο πρώτος. Ένα λεπτό κάθε μιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Φέρε Βάλντερ, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπε η Επίτροπος, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία στρατιωτική λύση, αυτό θα πρέπει να είναι πηχαίος τίτλος ε, στη Σρι ότι τα προβλήματα, οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά από πολλά χρόνια κατά βάση προσπαθεί η κυβέρνηση να τα επιλύσει, αλλά αυτό νομίζω αποτυχάνει λόγω της στρατηγικής επικοινωνίας και θα πρέπει επίση να δούμε ότι η στρατηγική θέση της Σρι κινητοποιεί δυνάμεις ε, διεθνώς που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν τοπικά. Θα πρέπει επίσης νομίζω να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και την οικονομική κατάσταση καλύτερα στα χέρια μας, να βελτιώσουμε τις υποδομές συγγνώμη, για να μπορεί να υπάρχει και ε, ενδυνάμει μια επικοινωνία μεταξύ των αντιμαχωμένων μερών, για να βρεθεί και λύση και έτσι. Ο κύριος Μάγερ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σρι ήταν ε, κάτι που μπορούσαμε να προβλέψουμε εδώ και κανένα δύο χρόνια. Δεν πρόκειται μόνο για ανθρωπιστικό πρόβλημα, αλλά πρόκειται και για μια πολύ σοβαρή πολιτική ε, σύγκρουση. Εδώ και χρόνια Ε, προσπαθούσε η κυβέρνηση να κάνει το διαμεσολαβητή ε, μεταξύ των, ε, της κυβέρνησης και των Ταμούλ. Ο Νορβηγός διαμεσολαβητής έκατσε αρκετά χρόνια αλλά κάποια στιγμή καταλήφθηκε η λύση της ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων. Η Σιριλάνκα έπαψε να προσπαθεί να βρει μια ειρηνική λύση και πέρασε σε μια μονομερή στρατιωτική λύση ναι. πλέον. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε δύο λαούς ε, οι οποίοι ε, τείνουν να απομακρύνονται ακόμα και περισσότερο, όλο και περισσότερο και η δυνατότητα συνεννόησης είναι όλο και πιο δύσκολη. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο και στο τέλος δεν θα υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ιτημένοι. Όλοι θα χάσουν. Ο κύριος Γκάλερ. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτρόπο για τα ανοιχτά της λόγια. Θα πρέπει νομίζω τώρα να στραφούμε στην μοίρα του αμάχου πληθυσμού και θα πρέπει να γίνει μόνο αυτό που είπε ε, στις 13 Δευτέρου το Συμβούλιο των Υπουργών, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή άμεση καταπαύση του, του πυρός. Δεν θα πρέπει να συμπληρώσουμε προσωρινό. Άμεση θα πούμε, αλλιώ η ανθρωπιστική καταστροφή στην οποία αναφερθήκατε θα συνεχιστεί. Και θεωρώ στην κατάσταση αυτή, στην οποία βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι εγκλωβισμένοι σε αυτή τη ζώνη και θέλουν να φύγουν από εκεί, θα πρέπει να είμαστε κατά οποιασδήποτε πράξη βίας που θα τους παρεμποδίζει από το να βγουν. Εμένα δεν, με ενδιαφέρει αν πρόκειται για τους τίγρε ή για τους στρατιώτες της κυβέρνησης. Εμένα με ενδιαφέρει ότι στρέφονται κατά τον άμαχον πληθυσμό. Εγώ θα ήθελα να στραφώ προς εκείνους ε, της ε, τέως απικιακής, ε, απικιοκρατικής δύναμης που φεύγουν αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα πρέπει να πιέζουμε μόνο τους τίγρες τα μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συζήτηση εδώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Εκτός ε, μικροφώνου κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι διαδικαστικό. Ήθελα απλώς να μιλήσω και εγώ στο κάτι Νόμιζα ότι το είχα καταφέρει, μου επιτρέπετε άλλωστε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, ήθελα απλώς εκτός ε, μικροφώνου το σχόλιο. Ναι, όντως ο πρόεδρος με είδε, αυτό επιτρέπεται. Ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μάγερ για τις παρατηρήσεις του αναφέρθηκε στην πολύτιμη δουλειά του κυρίου Ριξόλου από την Νορβηγία, τον οποίο συνάντησα προσφάτως στο Όσλο. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους συναδέλφους που μίλησαν με πάρα πολύ λογική. Όντως με τον άμαχο πληθυσμό ενδιαφερόμαστε και να σας επιστήσω την προσοχή συνάδελφοι από ότι όλες τις τροπολογίες η τροπολογία ένα είναι η πιο σημαντική η οποία ζητεί άμεση εκεχηρία που θα πρέπει να είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ιρλάνκα. Κάποια πράγματα δεν είναι απλά τυχαία. Είναι από την ε, Υπηρεσία Υγείας της ε, κυβέρνησης του Σρι Λάνκα και αναφέρεται σε ανθρώπινη καταστροφή και για τις επονίδιστες συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι στη Σρι Λάνκα. Αυτά τα υποστηρίζουν διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επομένως, ο όλος τίτλος αυτής της συζήτησης είναι η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα. Και εμείς έχουμε καθήκον να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τους συνδράμουμε και νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος δρόμος προς τα μπρο. Ευχαριστώ. Εγώ εφάρμοσα αυστηρά τον κανονισμό. Μπορούσαμε να ακούσουμε πέντε ομιλητές κατά τη διαδικασία και επομένω επειδή υπήρχε ακόμα δυνατότητα για επιπλέον ομιλητές έδωσα το λόγο στο συνάδελφο. Παρακαλώ η Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ του βουλευτέ για τη συζήτηση αυτή. Ήταν σύντομη συζήτηση, αργά τη νύχτα, παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι από την αρχή τη ε, Επιτροπή αυτή, ω συμπρόεδρο, ανησυχούσα πάρα πολύ για τη Σρι Λάγκα. Υπήρχαν στιγμέ όπου υπήρχαν ελπίδε, στην αρχή κυρίω, αλλά η ελπίδα αυτή εξαφανίστηκε. Υπήρχε η διαδικασία τη Γενέβη, την οποία επίση προσωπικά θέλησα να είμαι παρούσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο φαίνεται για την κυβέρνηση της Ριλάνκα. Δυστυχώς, οπωσδήποτε, αυτή η διδεξία δεν καρποφόρεσε Ήμουν έτοιμη να πάω και στον Βορρά για να αρχίσω ε, κάποια διαδικασία ε, διαμεσολάβησης, όπως ε, το είχε αρχίσει και ο Κρυς Πάτερ, ο προκατοχός μου. Αλλά δυστυχώς ο κ. Μπαζακαρά είχε, δεν ξέρω, αν φιλογιά κάτι τέτοιο. Συμφωνώ με τον κύριο Γκάλερτ που είπε, και αυτή είναι και η δική μου ανησυχία, ότι πρέπει πρώτα να βάλουμε τους ανθρώπους, πρώτα να ε, ενισχύσουμε την ανθρωπιστική πλευρά. Και πολλές φορές είμαστε οι μεγαλύτεροι ανθρωπιστικοί δότες στην Ευρώπη. 90 εκατομμύρια ε, δώσαμε το 2008-2009 για ανθρωπιστική ενίσχυση, το οποίο πέρασε από εταιρούς όπως το ε, Διεθνή στο Σταυρό, τα Ηνωμένα Έθνη και κάποιε διακυβερνητικέ οργανώσει. Αυτές οι οργανώσει ε, είναι έτοιμε να βοηθήσουν τον ε, πληθέντα πληθυσμό, αλλά έχουν προβλήματα πρόσβασης σε εκείνη την περιοχή. Από το Σεπτέμβριο του 2008, ο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό ήταν ο μόνος οργανισμό που επετράπη να ε, δράση στις ε, περιοχές που ελέγχονται από τους Σταμόλου. Καμιά φορά μπορέσαμε να στείλουμε κάποια τρόφιμα που κάλυψαν μόνο 50% των αναγκών. Δώσαμε επίσης άλλα σε 70 ε, εκατομμύρια ανθρωπιστικής βοήθειας στις διοργανώσεις το 2008 και ενισχύτη προσπαθούμε και σε επίπεδο Κολόμπο και σε επίπεδο Βρυξελών για καλύτερη πρόσβαση στις ε, ε, ε, ομάδες αυτές του πληθυσμού από κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι μαζί με τους άλλους συμπροέδρους, ιδίως με την Ολβηγία, εκμελευτήκαμε κάθε ευκαιρία που υπήρχε για να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την Συμφωνία κατάπαυση του Πυρός του 2002 και να επιλύσουμε την, λύση, την κατάσταση ε, ειρηνικά. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και όλες οι εγκλήσεις για την ε, επανάληψη των διαπραγματεύσεων δυστυχώς αγνοήθηκαν. Και έτσι η, η υπομονή της διεθνούς κοινότητας ε, μειώνεται. Κανένας όμως από τους συμπροεδρούς δεν έχει εγκαταλείψει το έργο του. Παραμένουμε προσκολλημένοι στην συμβολή μας σε μια ειρηνική επίλυση της διαμάχης όπως φαίνεται από την τελευταία δήλωση των συμπροεδρών της 3ης Φεβρουαρίου που είμαι σίγουρη ότι όλοι τη γνωρίζετε. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για ανθρωπιστική πρόσβαση να μπορέσουμε να βγάλουμε από εκεί, να ε, βοηθήσουμε να διαφύγει ο άμοχος πληθυσμός και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε ένα πολιτικό διάλογο με τα αντιμαχόμενα μέρη προσπαθώντας να τους πείσουμε ότι μόνο η πολιτική λύση είναι εκείνη που θα είναι μια λύση. Αλλιώς θα έχουμε ε, ανταρτοπόλεμο και αυτό δεν θα δώσει ποτέ την λύση πάνω σε αυτό το τόσο όμορφο νησί που ήταν παράδοσος και θα μπορούσε να ξαναγίνει παράδοση. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο για την παρουσία της και για τις παρεμβάσεις της στη συζήτηση. Η ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο ψηφίσματος θα γίνει αύριο στη συνήθεια ώρα των ψηφοφοριών. Οι εργασίες θα συνεχίσουν αύριο 10 με 1. Α, όχι, 9 με 1, 9 με 1, έκανα λάθος. Και κατόπιν μετά τις 3 το απόγευμα.